Pan Przewodniczący! Good morning. Please, please take a seat. Καλημέρα. Καθίστε. Παρακαλώ. Ας ξεκινήσουμε. Ξεκινήσουμε λοιπόν με κάποιες ε, πληροφορίες για τις πλημμύρες στην Ευρώπη. Υποφέρει και πάλι η Ευρώπη από πλημμύρες. Υπέφεραν περισσότερο το Βέλγιο, η Ολλανδία, η Ιταλία. Αυτή τη στιγμή έχουμε πλημμύρες στην κεντρική Ιταλία, στην νοτιοδυτική Ιταλία και σε άλλες χώρες. Ίσως όταν θα μιλήσω. Και αφού σας δώσω τον λόγο θα μας δώσετε και άλλα παραδείγματα. Υπήρχαν ε, νεκροί και ζημιές εκατομμυρίων. Και ξέρετε πως ε, πριν από 8 χρόνια συστάθηκε το Ταμείο Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν χρησιμοποιηθεί οι πόροι τους σε 33 περιπτώσεις μετά από φυσικές ε, καταστροφές. Ε. Συλλογούμαθα λοιπόν τις οικογένειες ε, των θυμάτων και αυτούς οι οποίοι έχασαν τις περιουσίες τους στις πλημμύρες. Είναι δραματικά αυτά τα γεγονότα. Οπότε τώρα κυρίες και κύριοι θα ήθελα να δώσω τον λόγο τους ε, εκπροσώπους των πολιτικών ομάδων. Πρώτος, εξ ονόματος του ΕΛΚ. Σιλβέστρη τον λόγο. Κύριε Πρόεδρε, τι τελευταίε εβδομάδε πολύ σοβαρέ ε, βροχοπτώσει έχουν πλέξει διάφορε ε, ευρωπαϊκέ χώρε και έχουν γονατίσει του ε, εκεί πληθυσμού. Έχασαν τη ζωή του τέσσερι Βέλγοι στο, στο Μπραμπάντ και στην στη Δυτική Φλάνδρα.